να προσπαθήσω να απαντήσω όσο γινόταν πληρέστερα. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Commissaire. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για αυτή την ε, απάντηση. Ε, κλείνει εδώ η συζήτηση. Ευχαριστούμε τους πάντες. Περνάμε στην επόμενη συζήτηση που αφορά στην προφορική ερώτηση στην Κομισιόν για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης για τους αστέγους. Δίνω το λόγο στον, ε, στην εισηγήτρια Ντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τελικά ε, έχουμε σε αυτό το κοινοβούλιο μία συζήτηση για τους αστέγους. Γι' αυτό θα ήθελα καταρχάς ε, να αποτίσω φόρο τιμής σε όλες τις οργανώσεις που όλη τη χρονιά δουλεύουν για να μπορέσουν να δώσουν βοήθεια στους πιο ευαίσθητους από εμά τους αστέγους. Ε, αυτή η έλλειψη στέγης είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας είναι ε, μία από τις πιο λυπηρές καταστάσεις της ανθρωπίνης φύσης. Είναι μία αδικία που δεν μπορούμε να αντέξουμε και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο δρόμο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική πολιτική πρόληψη. Αντί να κοιτάμε τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους από το δρόμο είναι να βιαστούμε λιγάκι να θέσουμε τέλος στις εξώσεις ε, στην κερδοσκοπία των ακινήτων και έτσι, ώστε να μειωθεί ε, αυτή ε, η έλλειψη στέγης ε, και η ομάδα, η, εικόνα του αστέγου έχει γίνει πολύ πιο πολύπλοκη σήμερα και πιο σκληρή. Έχουμε όλο και περισσότερο νέους, γυναίκες, οικογένειες μεταναστών, φτωχούς εργαζομένους. Είναι πολύ αυτοί που βλέπουμε ε, πάνω στο δρόμο κατά γης, να στέκονται πάνω σε χαρτόνια το χειμώνα. Ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στα καταφύγια και σε διάφορα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό κάθε μέρα οι οργανώσεις κρούν τον κόδωνα κινδύνου. Ε, όμως η αδράνεια είναι ένα σκάνδαλο. Ήρθε λοιπόν η στιγμή τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ήρθε η στιγμή να θέσουμε ένα τέλος σε αυτή την ε, ε επονίδιστη κατάσταση. Θα πρέπει ε, λοιπόν ε, να βρούμε αιφόρες λύσεις εναντί αυτής της πραγματικότητας και να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους. Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη αλήθεια ε, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Ε, φαίνεται ότι οι άστεγοι έχουν φύγει από το κέντρο της πόλης, τους διώχνουν προς την περιφέρεια για να μην τους βλέπουν οι τουρίστες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν τους βλέπουμε δεν υφίστανται πλέον. Το πρόβλημα είναι εκεί και πρέπει να το λύσουμε σε μια χώρα που γνωρίζετε καλά κύριε Πρόεδρε, οι άστεγοι θεωρούνται κλιματίες. Ε, δεν μπορούν να κοιμούνται στο δρόμο γιατί θα πρέπει να πληρώσουν ε, πρόστιμο και τους ε, κυνηγούγα η αστυνομία στις, στους σταθμούς. Πρέπει λοιπόν να βρούμε χώρο για να τους υποδεχτούμε. Υπάρχουν ε, πτώσεις υποσχέσεις που δεν τηρούνται από την κυβέρνηση και γι' αυτό η διάσκεψη συνένεση ε, για του άστεγους ε, προσπαθεί να βρει ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα μέχρι το 2020. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να διευθυνθεί γύρω από πέντε μεγάλους στόχους. Ε, από τη μία την πρόληψη της έλλειψης στέγης, την συγκέντρωση των προσπαθειών στα πιο ε, σοβαρά προβλήματα, μια βελτίωση των υπηρεσιών ε, προς τους αστέγους ε, και μια επάρκεια της στέγης. Με συντονισμένες προσπάθειες περιφερειακές και εθνικές θα μπορέσουμε τελικά να έχουμε καλούς δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινωνική καινοτομία. Η στέγη θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα μιας επανένταξης στην κοινωνία να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τη στέγη. Κύριε Επίτροπε, πέρα από τις λέξεις υπάρχει η επίγουσα κατάσταση που επιζητά πράξεις. Δεν είναι οι άστεγοι ε, ε, θύματα, δεν πρέπει να περιμένουμε το χειμώνα ώστε να βλέπουμε τους ανθρώπους να, ε, να κοίτανται εκεί. Ε, θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στην έλλειψη στέγης και να βοηθήσουμε τους αστέγους. Ευχαριστούμε. Ε, ο, ο λόγος στον Επίτροπο. Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, δεδομένης της πίεσης και των ε, άσχημων συνθήκων στις οποίες ζουν ζει ο κόσμος, δεν είναι εντυπωσιακό ότι η φτώχεια όλο ένα και περισσότερο συζητιέται εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να δούμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι άστεγοι υπήρχαν και παλιότερα, μόνο που η κρίση επιδίνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη. Υπάρχουν, ωστόσο, υπάρχει ωστόσο και αυξανόμενη κατανόηση του τι χρειάζεται για την αντιμετώπιση. Τα κράτη-μέλη χρειάζεται να συνεχίσουν να αναπτύχουν εθνικά και περιφερειακά προγράμματα δράσης για να αντιμετωπίσουν του άστεγου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κοινή έκθεση του 2010 για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Φυσικά τα κρατη είναι υπεύθυνα για πολλά από, τα χρειά, όσα χρειάζονται να γίνουν, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κρατη στις προσπάθειές τους. Για παράδειγμα, βοηθώντας τη βελτίωση και κατανόηση των προβλημάτων καθώς και στην κατανόηση των πιθανών λύσεων στην εξέβριση καλύτερων μέσων για την ε, κατανόησή τους, τη μέτρησή τους και τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία θα πρέπει και μπορούν να κινητοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι άστεγοι. Το Περιφερειακό Ταμείο παρέχει χρήματα για στέγαση για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχει βοήθεια για την κοινωνική επανένταξη των αστέγων και για την στέγασή του, Μιλάμε το, είμαστε τώρα μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2013. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα, η χρηματοδότηση από το Ταμείο συνοχή για την επίτευξη των στόχων του 2020 και για την περιορισμό τη στόχη είναι ζωτικής σημασίας. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Συνένεση εντόπισε πιθανού διάβλου και τους ακολουθούμε για παράδειγμα για τη βελτίωση της γνώσης και της παρακολούθησης δίνοντας ε, ε, προσεγγίσεις για την στέγαση. Επίσης η δήλωση του Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπεριαστέγων τονίζει διάφορες προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένες της ανάγκης για καλύτερες στατιστικές. Η Κομισιόν δραστηριοποιείται λοιπόν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των αστέγων είναι πολύ σημαντική ε, υπόθεση για την ε, αντιμετώπιση της στόχιας μέσα στη στρατηγική του 2020 και καλύπτονται τομείς που στονίζονται και στην διάσκεψη συνένεσης. Ε, μόλις έχει ξεκινήσει μια νέα μελέτη για τη σχέση μεταξύ των αστέγων και των μεταναστών. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανάπτυξη δικτών σε συνεργασία με την Επιτροπή Περικοινωνικής ε, ε, ε, Πρόνοιας και θα θέλαμε οι συστάσεις μας να εφαρμόζονται ευρύτερα. Αυτό που έχει σημασία ωστόσο τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε την ενέργειά μας και τους πόρους μας ώστε να υλοποιήσουμε τα, τους στόχους που έχουμε εντοπίσει και όχι να εισάγουμε νέες διαδικασίες ή, ή οδηγίες με τη μορφή ομάδων υψηλού επίπεδου ή επιτροπών. Την περασμένη εβδομάδα ε, ήρθα σε επαφή με διάφορους φορείς για την αντιμετώπιση των αστέγων και δείχνουμε και, και, βλέπουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να δοθεί αρκετή προσοχή και ενέργεια. Ο διάλογος συνεχίζεται και θα πρέπει να ακολουθηθεί και από δράση. Ευχαριστώ, Πέτροπε. Τώρα έχουν τον λόγο οι ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων και, και, και πρώτα ο κύριος Ορή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. οι σοσιαλιστές συνάδελφοι υποφάσισαν να απευθυνθούν στην Κομισιόν με αυτό το ερώτημα και θέλουν και μία ε, πρόταση ψηφίσματος. Το κόμμα μας είναι, η ομάδα μας ε, θεωρεί ότι αυτό ε, είναι δικαιολογημένο και υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Η έλλειψη στέγης είναι ένα, μια ακραία μορφή της φτώχειας. Επίσης, είμαστε της άποψης ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα. Γι' αυτό ε, χρειάζεται μία προσέγγιση ε, κατάλληλη. Ε, Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στα κράτη-μέλη, αλλά και στις διάφορες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η έλλειψη στέγησης είναι η τελική κατάσταση της, ε, του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο άστεγος δεν έχει πλέον δουλειά. Όποιος δεν έχει δουλειά δεν έχει καμία πιθανότητα να βγει από αυτή την κατάσταση. Ε, και υπάρχουν και άλλα προβλήματα, ασθένειες, ε, σωματική κατάρρευση, πνευματική κατάρρευση, πράγματα τέτοια, όπως επίσης δημιουργία συμμοριών, εγκληματικών ομάδων κτλ. Όλα αυτά είναι θέματα ε, που τίθενται και χρειάζεται γι' αυτό ένα κοινωνικό δίκτυο, εκπαίδευση, γιατί για παράδειγμα σε διάφορα κράτη-μέλη έχουμε παραδειγμάτα επιτυχημένων προσπαθειών. Πρώτα απ' όλα Λοιπόν, θα έπρεπε να δούμε ε, ποιες είναι οι καλές πρακτικές, να τις ε, μελετήσουμε και να δούμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Εμείς από την πλευρά μας λοιπόν χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση και την υποστηρίζουμε. Ε, ο λόγος τώρα στην κυρία Μπέρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι η δεύτερη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινητοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα για να απευθυνθεί σε εσά σε σχέση με το θέμα των αστέγων. Το 2008 η κρίση μόλις είχε ε, και φτάνουμε στο 2011 με μια δήλωση που είχε δημιουργηθεί το 2010 και αναφέρει πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση να αντιμετωπίσουμε αυτό το σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτό το χώρο ε, που σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί χώρο πλούτου και, και πολιτισμού, οι άστεγοι ε, βρίσκονται σε κάθε πόλη. Κάθε μέρα η τοπική η αυτοδιοίκηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτούς τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων είτε στην Αθήνα, στο είτε στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Ελσίνκι. Μπορούμε εμείς σε μια Ευρώπη αλληλεγγύης να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους άστεγους αυτή είναι η πιο ε, ξεκάθαρη εκδήλωση της φτώχειας ε, και, της, ε, κοινωνική, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όταν έχουμε λοιπόν στόχους επάταξης της φτώχεια φτώχειας μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε αν είναι θέμα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέματα που υπάρχουν στη χάρτα των, ανθρωπίν, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα πρέπει να αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Γι' αυτό, κύριε Πίτροπε, ε, το Κολέγιο των Επιτρόπων θα πρέπει να κινητοποιήσει τα μέσα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή της, ε, ώστε το Σύμφωνο Σταθερότητας να μην οδηγήσει ε, στην τυφλή περικοπή όλων των χρηματοδοτήσεων που φτάνουν σε αυτόν τον πληθυσμό. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παραδειγματική δουλειά ε, σε κοινωνικό επίπεδο και για αυτούς ε, είναι σχεδόν αδύνατο πλέον να δουλέψουν όπως φάνηκε στη Γαλλία με την επαρέτηση του Ξαβιέ Νομαλή που έκανε, είχε μεγάλο απόϊχο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η Κομισιόν να, να, οδηγήσει, να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να μην εφαρμόζουν τους κανόνες ανταγωνισμού ε, στην κοινωνική στέγαση και να σταματήσει το θέμα των αστέγων να αποτελεί επίγον ζήτημα. Ευχαριστούμε η κυρία Λίν για τρία λεπτά. Παρόλο που η πάταξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι μία από τις ευκαιρίες των εθνικών κυβερνήσεων να δείξουν τη δράση του, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονίσει τι προσπάθειες αυτέ, ειδικότερα στο θέμα τη έλλειψης ε, στέγη που σχετίζεται με τη στρατηγική για το 2020. Δεν θέλουμε να επαναφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν πολλά, πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να συλλέξουμε αυτέ τι πληροφορίε και να τι διαδώσουμε πολύ πιο ευρέω από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί η Κομισιόν λοιπόν να, μας παραθέσει τα σχέδιά της σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει σχετικά με την ε, στρατηγική για την ε, έλλειψη στέγης όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών. Επίσης, πόσα στοιχεία υπάρχουν ήδη από τα κράτη-μέλη για τα αίτια της ε, έλλειψη στέγης. Ξέρουμε ότι 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν δικό τους χώρο στέγασης. Ε, γιατί γίνεται αυτό, γιατί το αλκοόλ, ε, κατά πόσο το αλκοόλ και τα ναρκωτικά συνεισφέρουν σε αυτό το πρόβλημα. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, από τους αστέγους το 40% έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, 49% με τα ναρκωτικά και 35% έχουν πνευματικά προβλήματα. πολλοί από αυτούς επίσης έχουν πάνω από ένα από αυτά τα προβλήματα, ε, συνδυασμένο το πρόβλημα του αλκοολισμού, των ναρκωτικών και, της, ε, και των ε, ψυχικών προβλημάτων. Πόσο, πόσο το κατανοεί αυτό το θέμα η Κομισιόν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, στο πρόγραμμα Daphne, ε, ε, για παράδειγμα, αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες. Υπάρχουν άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη βία στο σπίτι, που και αυτή οδηγεί στο να γίνει κανείς άστεγος. Αυτό λοιπόν που όλοι μας επιζητούμε εδώ είναι μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω απ' όλα χρειάζεται να γνωρίζουμε τι έχει ήδη γίνει και πώς μπορούμε να συνδράμουμε ε, στην ε, ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών πολιτικών που ε, θα ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να θέσουν μία προθεσμία μέχρι την οποία θα σταματήσουν να υπάρχουν άστεγοι. Όπως είπε και η Καρίμα Ντελή, υπήρξε ένα κείμενο ε, που εκδόθηκε το Δεκέμβρη πέρυσι. Η άστεγη δεν ήταν ποτέ μια πολιτική ε, προτεραιότητα, ούτε ένα δημοφιλές θέμα. Ίσως επειδή δεν υπάρχουν πολλοί ψήφοι που να διακυβεύονται. Πολλές ψήφοι που να διακυβεύονται. Ένα σημαντικό όμω ζήτημα ε, που θα πρέπει να ενώνει όλα τα κόμματα, όλους τους ανθρώπους, περιφερειακά, εθνικά, ε, τους ε, όσους χαράσουν πολιτική και πάνω απ' όλα όλους όσους υπήρξαν άστεγοι κάποια στιγμή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική για τους αστέους που πραγματικά θα δουλέψει, μια στρατηγική για το μέλλον. Ευχαριστούμε την κυρία Λίν και τώρα ο κύριος Ξαρνέκη για δύο λεπτά. Mam szczególny powód, και εγώ με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση, διότι το θέμα αυτό είναι άκρος ενδιαφέρον. Στην Κρακοβία, το 19ο αιώνα, ένας πρόγονός μου είχε δημιουργήσει καταβλισμούς για τους άστεγους ε, ήταν δηλαδή πολύ παλαιό το, το πρόβλημα, πολύ παλαιότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τότε το κράτος δεν ήξερε πώς να το αντιμετωπίσει. Βέβαια σήμερα θα μπορούσαμε να επαναλαμβάνουμε και να λέμε ότι το θέμα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ένωσης, αλλά νομίζω ότι για πολλούς λόγους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι προπομπός και να πιέσει τα κράτη-μέλη να συντονίσουν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Η κρίση κατέδειξε ότι, ότι δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Είναι μια κατάσταση πλημμυρίδας και το πρόβλημα όλο ένα και διονγκώνεται. Μιλήσαμε για κερδοσκοπία στην κτηματαγορά, μιλήσαμε για τον τραπεζικό τομέα, για τα δάνεια. Όλα αυτά μπορούν ε, να οδηγήσουν σε ολοένα και περισσότερους άστεγους, σε έλλειψη στέγης γενικότερα. Το θέμα είναι ευρύτερο δηλαδή. Αφορά την, ε, τον σύγχρονό μας πολιτισμό, την κοινωνία καταναλωτισμού που δημιουργεί μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε με μία φωνή όλοι και να τονίσουμε το, την ηθική μας υποχρέωση ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους α, αναγκεμένους, ο αριθμός των οποίων ολοένα και ε, διονγκούνται. Κυρία Φιγκερέδο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρόβλημα των αστέγων αποτελεί μια παράδεκτη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι απαιτούνται αποτελεσματικά μέτρα. Όπως είπαμε στις 16 Δεκεμβρίου το 2010 στην ανακοίνωσή μας, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό για να μην κοιμάται κανείς στους δρόμους και να βρούμε και τρόπους προσωρινής στέγης, αλλά αυτό μόνο για μία αναγκαία χρονική περίοδο πριν βρεθεί μόνιμη στέγη. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει μία στρατηγική για τους αστέγους και τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια των ε, εθνικών του στρατηγικών θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κοινοτικά κονδύλια έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο. Θα πρέπει όμως η συλλογιστική των αστέγων να ενταχθεί στους βασικούς πολιτικούς τομείς, ιδιαίτερα στον οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και κοινωνικό, έτσι ώστε να υπάρχουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες που να προβάλλουν την αξιοπρέπεια. Αν προβάλλουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές ε, λιτότητα και δεν προωθήσουμε τον κοινωνικό τομέα, τότε οι άνθρωποι δεν θα έχουν τις προϋποθέσεις για να βρουν στέγη και δεν θα βρίσκονται σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Δηλαδή από το ενίκιο μέχρι το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο, τη θέρμανση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το φαινόμενο των αστέγων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού μας και οι άνθρωποι που διαβιούν στο δρόμο είναι ύψη στη μορφή φτώχειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ε, πρόβλημα πολλές φορές όταν χάσει κανείς το σύντροφό του, όταν χρησιμοποιεί ναρκωτικά, όταν πρέπει να μεταβεί σε μια άλλη χώρα, όταν δεν έχει πια εισόδημα, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Με τη δήλωση μας πέρσι το Δεκέμβριο προσπαθήσαμε να βρούμε ενδεχόμενες λύσεις. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε το θέμα των εξώσεων, το οποίο θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε. Επίσης, ως προς την προσωρινή στέγη θα πρέπει να υπάρχει αρχικά, μέχρι κανείς να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα και οι άστεγοι στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε στέγη την οποία, τις οποίες το ενίκιο να μπορούν να καταβάλουν. Χρειάζονται πολλές μορφές βοήθειας οι άστεγοι, αλλά αυτό θα πρέπει να σημαίνει την, ε, δραστηριότητα, την άμεση δραστηριότητά τους. Ντότς για μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, Επίτροπε. Συνάδελφοι, εγώ καλωσορίζω την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση για το θέμα της έλλειψης ε, στέγης ε, και ενώ αναγνωρίζω ότι πρόκειται για ένα θέμα για τα κρατημέλη, είναι επίσης ένα θέμα που αυτό το κοινοβούλιο μπορεί να, δώσει, να του αποδώσει περισσότερη πολιτική σημασία μέσω τέτοιου είδους αναγνώρισης και τέτοιου είδους συζήτησης. Το 2010 και με 2011 στη δική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία, ο αριθμός των ανθρώπων που καταγράφηκαν ως άστεγοι αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το 2010 υπήρχαν πάνω από 38.000 υποψήφοι στο ε, λίστα αναμονής για κοινωνική στέγαση και βέβαια μεγαλύτερος αριθμός αστέγων αλλά και μεγαλύτερος αριθμός ετούντων κοινωνικής ε, στέγασης και αυτό το ακούσαμε για το, τους λόγους στους οφείλονται όλα αυτά. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι να δώσουμε επαρκή υποστήριξη, καθοδήγηση και κατάρτιση σε όσους τους βοηθούν ε, αλλά και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση καθώς και να τους προμηθεύσουμε προσιτή στέγαση. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες στη Βόρεια Ιρλανδία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αστέγων. Στα τελευταία τρία χρόνια 200 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για κοινωνική στέγαση και ενθαρρύνομαι ιδιαίτερα γιατί δίνεται έμφαση στους νέους ανθρώπους που βρίσκονται άστεγοι μένει με δύσκολα, προβλήματα, πολύ με δύσκολα προβλήματα και θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο χρόνο ξεκίνησε μια καλή πρωτοβουλία για να δοθούν στους νέους μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία μέσω της παροχής ε, κατάλληλης ε, στέγασης και στήριξης. Αυτά είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει όλοι να τα υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντότζη. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Σαγιά για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η άστεγη είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, στην Ευρώπη και είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα με το οποίο συνδέονται και άλλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τον αστέγους με ένα μοναδικό τρόπο, με έναν ενιαίο τρόπο γιατί το φαινόμενο διαφέρει από χώρα σε χώρα και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια κοινή πολιτική, ωστόσο αυτό θα μπορεί να αποτελέσει ε, δικαιολογία, πρόσχημα για την έλλειψη στρατηγικής. Θα πρέπει να ρυθμίζεται αυτό από τα κάτι μελη αλλά χρειάζεται ένα συντονισμός καθώς και ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών. Ε, είμαι ευτυχής που πολλές χώρες ωστόσο έχουν εθνικές στρατηγικές και στην χώρα μου έχουμε προγράμματα για τους μακροχρόνια αστεγούς και τον περιορισμό αυτών που από που, που, βασίζεται στην αρχή του στέχασης πρώτα. Δηλαδή, θέλουμε να, να δώσουμε κίνητρα σε όσους έχουν προβλήματα εξάρτησης από το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, ε, να προλάβουμε δηλαδή την ε, ε, έλλειψη στέγης και όχι να βασιστούμε μόνο στην κατασκευή προσωρινών κατοικιών. οι υπάρχουσες ε, τα, κατοικίες είναι φθηνότερες ε, για την αντιμετώπιση των αστέγων παρά η δημιουργία προσωρινών καταλήμματων ή η στέγασή τους σε νοσοκομεία ή φυλακές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τάρτα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως εισηγητής ε, για το θέμα της φτώχειας ε, και της κρίσης στα κράτη-μέλη. είμαι ότι μια οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν βασιστεί μόνο στην δημοσιονομική πειθαρχία. Η στόχοι της στρατηγικής 2020 είναι θεμελιώδης και ιδιαίτερα η μείωση της φτώχειας. Οι κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν να περάσουν σε δεύτερο πλάνο. Θα πρέπει να, να, να εφαρμόζονται παράλληλα με την δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να μειωθεί η φτώχεια και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις όπως η στήριξη της ευρωπαϊκής κατανάλωσης. Η ε, άστεγοι βεβαίως ε, για τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε φτώχεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό είναι το πιο προηγμένο στάδιο. Από τη στιγμή που έχουν αποκλειστεί από την αγορά απασχόλησης το άτομο έχει πρώτη του προτεραιότητα το που θα κοιμηθεί κάθε βράδυ και, και υποστηρίζω τα όσα προτείνονται στο προφορική ερώτηση και στην, στο ψήφισμα, δηλαδή η, δημιουργία προσιτών ε, κατοικιών. Η κοινωνική κατοικία είναι θέμα των κρατών μελών και είναι ελεύθερη, ελεύθερα να το προάγουν όπως δει. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να παρεμπαδιστούν στον αγώνα ε, κατά των ε, έλλειψη στέγης μέσω όσον αφορά τις, την βοήθεια που δίνουν και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα που ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία και έτσι να μπορώ να την παραθέσω στη μελλοντική μου έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος ο κύριο Μέρφη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν έγινε αναφορά στην, ε, στους στόχους του 2020 να βγουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια και την κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι τότε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως την πραγματικότητα. Αντί να προσεγγίζουμε το στόχο όλο και απομακρυνόμαστε από αυτόν. Και αυτό είναι άμεσο ε, αποτέλεσμα των επιθέσεων σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη. Αυτές οι πολιτικές ε, λιτότητας σπρώχνουν πολλούς στο να γίνουν άστεγοι. Στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια ε, οι άστεγοι έχουν αυξηθούν στην Ιρλανδία. Ε, ήταν αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό σημαίνει λιγότερη πόρη για την ε, κοινωνία μας ε, και υπάρχουν και χειρότερες συνθήκες για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Ε, αυτές οι επιθέσεις που βασίζονται στο κέρδος και όχι στις ανάγκες των ανθρώπων έχουν βάλει 48.000 οικογένειες στην Ιρλανδία στις λίστες αναμονής. Ε, κανείς ακόμα δεν έχει αποφελθεί από τα χρήματα που δίνονται ε, βασίζονται όλοι στον ιδιωτικό τομέα και μόνο ε, ε λίγες ήταν οι στέγες που εξασφαλίστηκαν ε, στην Ιρλανδία για τους αστέγους. Όμως οι τραπεζίτες και είναι αυτοί που ζητούν περισσότερα χρήματα και δεν δίνονται πλέον αυτά στους αστέγους. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να βρουν ε, ο κόσμος στέγη ε, άμεσα. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στην κυρία Ντελβό για δύο λεπτά. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για αυτό το ψήφισμα για την έλλειψη στέγηση γιατί μας θυμίζει την ευθύνη μας να αντιμετωπίσουμε την επίγουσα αυτή κατάσταση. Αυτό που χθες ήταν προτεραιότητα σήμερα είναι ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη. Υπάρχουν κάποιοι ε, δεν υπάρχουν ε, ε, δείκτες αξιόπιστοι, όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να διαπιστώσουμε ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί. Έχουμε φτάσει στα 84 εκατομμύρια το 2011 σύμφωνα με τη Eurostat. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία θα ήταν σωστό να τεθεί ένα τέλος αυτό το πρόβλημα μέχρι το 2015 σύμφωνα με τη στρατηγική. Ελάχιστα έχουμε προσεγγίσει αυτό τον στόχο. Το 2010 ήταν ε, το έτος κατά της φτώχειας και το χρησιμοποίησαν ε, τα κράτη-μέλη ε, και τελικά το για να κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο σταθερό. Ε, το, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει μια ε, παγκόσμια πολιτομεακή πολιτική για την έλλειψη στέχης, ε, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για θέματα οικογενειακά, θέματα υγείας και θέματα προσωπικής ευπάθειας που συνδυάζονται με την έλλειψη στέχης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική πορεία του κάθε αστέγου για να μπορέσουν ε, να, ε, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τικάου. Ε, μια ερώτηση. Ε, ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση προς τη συνάδελφο. Εγώ άκουσα ότι 84 εκατομμύρια είναι άστεγοι. Καλά άκουσα ή δεν άκουσα καλά. sunt expuși riscului sărăciei, dar nu Δηλαδή, ίσως εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας, αλλά όχι ότι είναι άστεγοι. Non, madame, à mon avis, c'est Αλλά είναι πρόβλημα μετάφραση, γιατί είναι αυτοί που έφτασαν ε, κάτω από το κατόφλι τη ε, ε, φτώχεια. Ναι, όντω ήταν σωστή η ερώτησή σα. Ενδιαφέρει του πάντε. Περνάμε στην κυρία Γκάγκ για τρία λεπτά. Ε, ευχαριστώ. Να θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, δραστηριοποιηθεί σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με το συντονισμό της στρατηγικής για, την, για τους αστέγους. Και με την διάσκεψη συνένεσης για την έλλειψη στέγης. Υπάρχουν και νέα φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει στο να χάσουν ε, για πολύ καιρό τη δουλειά τους ε, πολλοί άνθρωποι και πολλοί οικογένειες να μην μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα, ειδικότερα για αυτούς που πρέπει να πληρώσουν δάνεια σε συναλλαγμα. Ας πούμε σε, στο ελβετικό νόμισμα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν πολύ σημαντικά μέτρα. Για παράδειγμα, η οδηγία ε, που αφορά στην προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να φροντίσει για αυτό το θέμα. Όσον αφορά επίσης τις διακρίσεις κατά των αστέγων, Ε, που για πολλές, σε πολλές περιπτώσεις διώκονται και πρέπει να πληρώσουν και πρόστιμα. Η έλλειψη στέγης είναι μια ακραία μορφή της φτώχειας όπως είπαμε και θα πρέπει να αφιασιωθούμε ε, πιο πολύ σε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μέγερ για 1,5 λεπτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα περιορίζοντας το κόστος, διότι αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει ευεργέτημα των εχόντων ανάγκη και των αστέγων και αυτό το είδαμε και στις ΕΠΑ. Το θέμα της αντιμετώπισης των αστέγων δεν αντιμετωπίζεται το θέμα με καλές προθέσεις θέσεις. Ίσως εμάς στην Ιταλία μας πλήττει η ανεργία πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Υπάρχουν πολλοί άνεργοι, ε, άνθρωποι που πρέπει να καταβάλουν κάθε μήνα ε, το δάνειό τους, τη δόση του δανείου. Και πρέπει με κάθε τρόπο να το κάνουν. Είτε έχουν είτε δεν έχουν εισοδήματα. Αυτό είναι ανήθικο. Γιατί θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί τι γίνεται, γίνονται και κατασχέσεις οικειών στην περίπτωση που κανείς δεν μπορεί να καταβάλει τη δόση του δανείου. Αυτό είναι ανήθικο, θα πρέπει τη στιγμή που κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του δανείου, δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος να ε, ε, καταβάλει μία δόση ενός ε, δανείου τη στιγμή που δεν διαθέτει κανένα εισόδημα. Αυτό είναι καθαρά ανήθικο και θα πρέπει να αλλάξουμε αυτόν τον ε, οικονομικό προσανατολισμό που είναι καθαρά φιλελεύθερος. Η κυρία Σριντένσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα των αστέγων δεν έχει επιληθεί στην Ευρώπη οι άστεγοι αλλάζουν χαρακτηριστικά. Συνήθως είχαμε την εικόνα ενός μεσήλικα ο οποίος κοιμάται στο δρόμο. Έχουμε όμως και νέες γυναίκες ή μετανάστες ή θύματα βίας που δεν έχουν στέγη. Το θέμα λοιπόν των αστέγων αφορά την, το γεγονό ότι δεν διαθέτει κανείς στέγη και ότι πρέπει να κοιμηθεί στο δρόμο. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίε στα κράτη-μέλη, καθώς και η μεθοδολογία ομοσυλλογής στοιχείων διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε την κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταπολεμήσουμε την ε, μη διάθεση στέγης. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποβάλω ορισμένε ερωτήσεις. Πέρσι το Δεκέμβριο έγινε μία διάσκεψη συνένεσης για τους αστέγους και υπήρξε διαφοροποίηση, κατηγοριοποίηση δηλαδή λόγων που οδηγούν στην έλλειψη στέγης. Τι θα κάνουμε, θα συμπεριλάβουμε αυτές τις διαφορές, θα τις συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προβάλλει διαφορετικά μέτρα ανάλογα με τους λόγους έλλειψη στέγης. Θα συμμετέχουν και οι ΜΚΟ σε αυτή τη διαδικασία. Και πώς θα συμμετάσχουν έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η έλλειψη στέγης. Επίσης, τη στιγμή που θα εφαρμοστεί η στρατηγική, πώς ε, θα είναι πραγματικά αποτελεσματική τη στιγμή που έχει διαφορετικό ε, πρόσωπο σε κάθε χώρα. Η κυρία Μπένοβα. Κύριε Επίτροπε, το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο Ρώτησα την Επιτροπή με τους άλλους συναδέλφους κατά πόσο προβλέπεται μία στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αστέγων. Δραστικά τι έχει γίνει έκτοτε, ποια μέτρα ελήφθησαν και θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας στην εκπόνηση αυτής της στρατηγικής για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αστέγων, των αστέγων που κοιμούνται στους δρόμους. Θα πρέπει να είναι μία στοχοθετημένη πολιτική η οποία να έχει σαφείς διαστάσεις και να λάβει υπόψη τα διάφορα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ολοένα και διουγκούμενη φτώχεια στα κράτη-μέλη. Η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση των αστέγων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα εθνικά σχέδια και εθνικά προγράμματα συντονισμού για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ποια είναι τα μέτρα λοιπόν και τι προβλέπετε για να συνεργαστείτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βερζιά, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 8% των Ευρωπαίων ζουν σε μια κατάσταση ένδυας και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές τους ανάγκες. Πολλοί ζουν στους δρόμους ή σε προσωρινή στέγη, η οποία δεν ε, προϋποθέτει συνθήκες υγιεινής. Αυτό αφορά γυναίκες, παιδιά, μετανάστες και δεν μπορούν να ζήσουν μια σωστή η οικογενειακή ζωή. Βεβαίω η κρίση επιδίνωσε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν η πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Οι πολιτικές λιτότητα πλήττουν τους πλέον ενδεεί. Δεν έχουμε πλέον τα κατάλληλα μέσα. Και πέρα από τα μεγάλα λόγια, ποιες είναι οι ουσιαστικές πολιτικές των κρατών μελών τη στιγμή που δεν μπορούν να μας δώσουν ούτε στατιστικές επί του θέματος. Ακόμα χειρότερα, Δυστυχώς ορισμένα κράτη-μέλη ποινικοποιούν τους άστεγους την κατάσταση αυτή. Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τους πλέον φτωχούς. Δεν έχουν νόημα τα παχιά λόγια για τα δικαιώματα του, του ανθρώπου και την κοινωνική πρόνοια. Η κυρία Μπάστος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο αριθμός των αστέγων, όπως και των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της στόχης, δεν ε, σταματά να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη. Η κρίση οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική και η αύξηση της ανεργίας επιδίνωσαν αυτό το πρόβλημα, όπως όλοι ήδη ανέφεραν. Επίσης όλοι συμφωνούμε πως αυτό το φαινόμενο είναι η αρνησή σημαντικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο σεβασμός στην ανθρώπινη εξωπρέπεια και ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή υπόκειται σε πολύ αυστηρά μέτρα λιτότητας, έννοια του αστέγου συμπεριλαμβάνει και τους ανθρώπους που δεν μπορούν και αναζητούν βοήθεια για να μπορέσουν να φάνε και ο αριθμός αυτών αυξήθηκε κατά 20% από το 2008 οικογένειες και άνθρωποι που είδαν να αναλάζει η κατάσταση της ζωής τους λόγω της ανεργίας και λόγω της ε, χρέωσής τους ε, στις τράπεζες. Ε, επιδεινώνεται η κατάσταση το περασμένο χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω μιας γραπτής δήλωσης για στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αστέγους τόνισε την ανάγκη να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια στρατηγική που θα αποτελείται από εθνικές και περιφερειακές ε, πολιτικές για μια μακρόπνοη στρατηγική για τους ανθρώπους που ζουν στο δρόμο, που κοιμούνται στο δρόμο. Θα πρέπει να υπάρξουν προληπτικά μέτρα αλλά και συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των αστέγων και για την δημιουργία προσιτών κατοικιών. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική οφείλει να είναι συμβατή με την πολιτική κοινωνική στέγαση των κρατών μελών. Καταγράφουμε λοιπόν τα λόγια του Επιτρόπου και τις προτάσει που μα έκανε. Περιμένουμε και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει σαφή και στεναρή όθηση ώστε να αναγκαστούν τα κράτη-μέλη και να, να καταπολεμήσουν αυτή την κοινωνική αδικία. Σα ευχαριστώ <coughs> κυρία Μπάστο, Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κοτσολίνο για 1,5 λεπτό. Α, είναι παλά. Είναι παλά λείπει. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, Μέντες Δεβίγκου, για δύο λεπτά. Ah, Στο τσακ, κύριε Μέντες. Πηγαίνετε αλλού. Και γρήγορα, κύριε Μέντες. C'est votre doigt, mon avis. Hein? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και το 2008 έγινε, το 2010 ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και είχαμε υποβάλει μία προφορική ερώτηση στην Κομισιόν. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ε, ανησυχεί για αυτήν την κατάσταση γιατί είναι πραγματικό το πρόβλημα. Πολλές φορές ε, ε, λέγεται ότι ασχολούμαστε με θεσμικά ζητήματα που δεν απασχολούν τον κόσμο. Δείχνουμε όμως ότι ανησυχούμε για θέματα και ζητήματα που είναι ουσιαστικά και πραγματικά. Είπε ο Επίτροπος ότι τα προγράμματα δράσεις είναι εθνικά προγράμματα. Αυτό είναι γεγονός. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το είπε και η κυρία Μπερές, διότι στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων μιλήσαμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό και θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Νομίζω ότι πολύ σύντομα και πολύ άμεσα μπορούμε κάτι να κάνουμε. Μιλώ για το, την ψήφιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημοσιονομικών μας προοπτικών. Επίσης, Πρόεδρε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια και οι άνθρωποι να έχουν την αξιοπρέπειά τους. Όποιος είναι φτωχός είναι ένας άνθρωπος που έχει όλα τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα. Ε, θα ήθελα να δείτε το φιλμ για τον πατέρα Περσίνσκι, ο οποίος ε, καταπολεμεί τις ε, ανισότητες αυτές. Φαίνεται ότι μας ενδιαφέρει να προωθούμε το δικό μας οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο. Αλλά αυτό δεν αφορά μία πολιτική ομάδα αφορά θέμα ουσίας και ταυτότητας, ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να ακολουθούμε πάντα αυτή την πορεία. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία κύριε Επίτροπο, ξέρετε, ένας άνθρωπος όσο φτωχός και να είναι, όταν περπατάει στο δρόμο και βλέπει έναν άστεγο, νομίζει ότι έχει τεράστια απόσταση από αυτόν κανένας φτωχός άνθρωπος δεν έχει στο μυαλό του ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει άστεγος κι όμως η διαφορά είναι ελάχιστη είναι μία τρίχα και αυτό αποδεικνύεται σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Η ρυθμοί αύξησης των αστέγων είναι μεγάλη. το νιώθουμε και χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα γιατί δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία όμως ο καθένας στη χώρα του στον τόπο του στη γειτονιά του ξέρει τι συμβαίνει και βλέπει τι συμβαίνει. όταν υπάρχει οικονομική κρίση υπάρχει φτώχεια. όταν υπάρχει φτώχεια σιγά σιγά έρχεται η έλλειψη απασχόλησης και εργασίας και ξαφνικά μέσα σε εισαγωγικά ένας άνθρωπος γίνεται άστεγος. αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και, όχι μόνο κάθε κράτος μέλος χωριστά. χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική μια ευρωπαϊκή ομπρέλα για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που κατ' εμέ θα πρέπει να είναι η κοινωνική επανένταξη των αστέγων. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ράπτη. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σαχτιέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτή την προφορική ερώτηση και αυτό το ψήφισμα διότι βρισκόμαστε ενώπιον ενός αναξιοπρεπούς προβλήματος. Αν είναι αναξιοπρεπές ε, για την ε, Ευρώπη, για τις αξίες που υποστηρίζουμε και για τα μέσα που έχουμε σε επίπεδο της Ευρώπης. Η κρίση επιδίνωσε και τόνισε το πρόβλημα των αστέγων. Πιστεύω όμως πως σήμερα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως όλοι μπορούν, μπορεί να πέσουν σε αυτή την παγίδα. Ναι, Οποιοδήποτε Ευρωπαίος μπορεί να βρεθεί άστεγος από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρώτο σημείο στο οποίο μπορούμε να ενεργήσουμε είναι βεβαίω το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που επιτρέπει την ένταξη, την επανένταξη στον ε, κόσμο της απασχόλησης, ε, προσαρμογή σε νέες θέσεις απασχόλησης, επιστροφή του ανέργου στην απασχόληση. Αλλά πέρα από αυτό, ως πρόεδρος εργασίας, ε, της ομάδας εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Progress, θα ήθελα να τονίσω το πρόγραμμα Progress μπορεί επίσης να μας βοηθήσει και οφείλει να μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην επίλυση του προβλήματος. Πρόληψη αλλά και καθορισμός από κοινού δικτών για να έχουμε μια πραγματική πολιτική με αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόσβαση στην στέγαση. Υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλές πρακτικές για την επίτευξη αυτών των στόχων. Πιστεύω πως όλοι μαζί οφείλουμε σε επίπεδο της Κομισιόν και στο επίπεδο της ομάδας εργασίας μας στην Επιτροπή ε, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την Πρόεδρό μας κυρία Μπερές να δούμε τι λειτουργεί στα κρατημέλη, ποιες είναι οι, πραγματικά, οι στρατηγικές μάλλον που έχουν μέλλον και αν πραγματικά ε, η προσωπική η ατομική προσέγγιση και η προσωπική παρακολούθηση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, το οποίο όπως σας είπα δεν είναι άξιο ε, είναι αναξιοπρεπές για την Ευρώπη. Ευχαριστώ, κυρία Τικάου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το θέμα των αστέγων δεν έχει μόνο ευρωπαϊκή διάσταση. Αφορά και το θέμα της ε, στέγης αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα το χειμώνα το πρόβλημα οξύνεται και υπάρχουν προσωρινέ, υπάρχει προσωρινή στέγη για τους αστέγους. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να βρούμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του αποκλεισμού ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό θα πρέπει να συντονιστούν οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως το θέμα διαφέρει μεταξύ κρατών μελών και αυτό αφορά και τη συλλογή στοιχείων και τη μεθοδολογία συλλογή στοιχείων. Θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό πλαίσιο για την κατάρτιση πολιτικών έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των στέγων για όλες τις εποχές και για πάντα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις πιο ευάλωτες κατηγορίες, δηλαδή τους νέους, ε, τους άνερους, πολύ μεγάλους, τα παιδιά, τους μετανάστες και να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στις πλέον μειονεκτικές περιχέρειες που πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του ΕΤΠΑ έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες. Το λόγο. Ευχαριστώ λόγο ε, στον κύριο Σόνικ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ένας από τους πέντε στόχους ε, της ε, Στρατηγικής Ευρώπης 2020 ε, είναι η άρση της φτώχειας για 20 εκατομμύρια ανθρώπους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στατιστικά στοιχεία του 2009 σχετικά με τη φτώχεια είναι ανησυχητικά. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους ε, που ζουν ε, στο όριο της φτώχειας και είναι κοντά στο να μείνουν άστεγοι. Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης. Η έλλειψη στέγης είναι ένα, μια δραματική πτυχή της φτώχειας ε, και μέσα από τις γενιές ε, βλέπουμε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να την πατάξουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να πατάξει το φαινόμενο αυτό. Έχουμε κάνει έκκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να πατάξουν την έλλειψη στέγης, ειδικότερα τους άστεγους που βρίσκονται στους δρόμους μέχρι το 2015. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα έντια αυτής της, αυτού του φαινομένου μέσα από σωστές στρατηγικές έβρεση στέγης. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι στην στρατηγική μας ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρέπει να κινητοποιήσει τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ετοιμάσουν και να σχεδιάσουν κατάλληλες στρατηγικές που θα ε, εκριζώσουν την έλλειψη στέγης. Επίσης πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία ε, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην εκκριζώση του προβλήματος, θα πρέπει ε, να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας ε, και τα διάφορα προσκόμματα. Πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να εφαρμόσουμε μέτρα που ίσως δεν είναι γραμμένα στο ε, νόμο, να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ εν τη ενώση. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Σμόλκοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Πίτροπε. Η άστεγη είναι μία από τις πιο ακραίες και χειρότερες μορφές ε, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καθημερινά συναντούμε αστέγους ε, μπροστά στα πολυκαταστήματα, ε, στις υπόγειες διαβάσεις. Βλέπουμε ε, πεινασμένους και βρώμικους ανθρώπους πολύ συχνά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα για μια αξιοπρεπή ζωή. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι μια κοινωνία ε, εποφελείται από την ε, πάταξη της φτώχειας. Γι' αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουν και να δραστηριοποιηθούν όλοι οι τομείς μιας κοινωνίας και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός ε, οι εκστρατείες ευαισθητοποίηση έχουν ε, μεν σχεδιαστεί, αλλά τώρα ε, ήρθε η στιγμή να φτιάξουμε και ένα σύστημα συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε την κυρία Σμόλκοβα. Περνάμε στη διαδικασία Κατστιάη, ο κύριος Νικολάζη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, πολλές φορές ε, βλέπουμε ε, ανθρώπους άστεγους οι οποίοι έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση λόγω πολλών αιτιών και αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Οι προσπάθειε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να επικεντρωθούν στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να δημιουργήσουν στέγη, δυνατότητε στέγαση για τους ε, φτωχού. και μεταξύ των άλλων θα πρέπει να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τους ε, αστέγους τα οποία θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται. Έλλειψη στέγης δεν μπορεί να γίνει κατανοητή εύκολα ε, σε μια ε, σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία το πρέπει να αποτελεί κομμάτι της. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα 20 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα πρόθυρα αυτής της κατάστασης. Ο κύριος Νικολάτσικη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρόβλημα των αστέγων είναι αδιαφυσβήτητα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όμως θα πρέπει να μην αγνοούμε κι άλλο ένα πρόβλημα ε, που είναι το ίδιο σοβαρό, την επισφαλή ε, κατάσταση ε, στις, τις συνθήκες διαβίωσης για κάποιους ανθρώπους που ζουν χωρίς ε, τουαλέτα, χωρίς ε, να, έχουν, ε, να κάνουν ένα μπάνιο. Πάνω από 8 εκατομμύρια Γάλλοι, για παράδειγμα, ζουν σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει, λοιπόν, πέρα λοιπόν από την πολιτική για τους αστέγους, θα πρέπει να έχουμε και μια μακροπρόθεσμη πολιτική για να βελτιώσουμε την κατάσταση διαβίωσης, τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων. Ο κύριος Λουάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόβλημα των αστέγων έχει γίνει πιο οξύ τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερες γυναίκες ε, γίνονται άστεγοι ε, και νέες οικογένειες, νέα παιδιά. Εργαζόμενοι που χάσαν τη δουλειά τους και μετά το σπίτι τους εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης να κάνω μελικέ προτάσεις στην Κομισιόν σχετικά με τι πιθανές λύσεις του προβλήματος. Καταρχάς θεωρώ ότι η δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Γραφείου για του αστέγους θα μπορούσε να αποτελέσει καλή ιδέα, διότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα και λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να διευρύνουμε τη χρήση των διευθυντικών ταμείων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να μπορέσουμε μια, να έχουμε μια καλύτερη ανάλυση του φαινομένου των αστέγων και ειδικότερα για να δημιουργήσουμε στέγη για τους αστέγους όπου χρειάζεται ε, επίσης ε, να γενικεύσουμε το φιλανδικό μοντέλο Και τέλος, ε, γιατί μειώνεται το κόστος, και τέλος θα πρέπει να βοηθήσουμε τους αστέγους και τις ενώσεις που τους υποστηρίζουν στη δημιουργία νέων μέτρων η κυρία Ζαβόρσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να πω ε, κάτι που δεν ακούστηκε σήμερα. Αν ε, ε, υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας, δεν υπάρχουν άστεγοι. Εμεί θα πρέπει να το έχουμε αυτό στο υπόψη μας. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώς υιοθετεί νομοθεσίες οι οποίες ε, αποδυναμώνουν την οικογένεια. Θα πρέπει οι μητέρες ε, να ε, μην έχουν πρόβλημα για τη φύλαξη των παιδιών τους. Αρνούμαστε στο Κοινοβούλιο να αναγνωρίσουμε την αξία μιας γυναίκας που φροντίζει το σπίτι της, την οικογένειά της, τους συγγενείς, τους γονείς της. Όταν βλέπουμε αστέγους, αμέσως προσπαθούμε να βρούμε στρατηγικές, να κάνουμε μελέτες και ξεχνάμε ότι η βάση όλων αυτών είναι η οικογένεια. Ευχαριστούμε την κυρία Ζαμπόσκα, κύριος Ματούλα για ένα λεπτό. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες ε, στέγης, διότι αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μειωθούν οι απόρριες αυτού του φαινομένου για να λάβουμε υπόψη την πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τους φτωχούς. Έχει μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε στέγη για εκείνους που χρειάζονται. Το ευρωπαϊκό έτος για την ε, αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις μπορούν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Θα ήθελα να μιλήσω και για συγκεκριμένες εθνικές στρατηγικές υπέρ των ευάλωτων ανθρώπων για την βελτίωση των συνθήκων ζωής, για την βελτίωση της ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και πρόνοιας, έτσι ώστε να, να υπάρχει προσβασιμότητα στη στέγη. Κυρία Πρέντεργκαστ. Ευχαριστώ. Να ερωτήσω, η Κομισιόν σκοπεύει να εξετάσει την χρήση κατοικιών που δεν, ε, που δεν κατοικήθηκαν ποτέ από την αρχή της κρίσης και έπειτα θα γίνουν προσπάθειες για ανακούφιση των οικονομικά πιεσμένων σπιτικών λόγω των τραπεζικών τους δανείων γιατί και αυτά αντιμετωπίζουν κίνδυνο να γίνουν άστεγοι. Και έπειτα υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ε, ε, πολοδομία, τον δανεισμό και την ανεργία για πολλά από αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό έχει διαφοροποιηθεί τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής κρίσης. Η έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής για την κοινωνική ολοκλήρωση και τη συμπερίληψη αυτών των, αυτής της κατηγορίας οδηγεί σε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα το θέμα των αστέγων έτσι ώστε να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή και πλήρη δικαιώματα. Να μην υπάρχει αυτός αποκλισμός διότι δημιουργεί ε, διακρίσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την φυσική και ψυχική ακαιρεότητα αυτών των ανθρώπων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχουν η συμμετοχή των κοινωνικών ταμείων και του ΕΤΠΑ έτσι ώστε να βρούμε μόνιμες μορφές στέγης. Και τέλος, το λόγο έχει ο κύριος Ανασέσκου. Ευχαριστώ. Από βιολογικής πλευράς η κατάσταση υγείας δεν είναι επανάκια ούτε προνόμιο των πλουσίων. Από κοινωνικής πλευράς όμως κάτι τέτοιο βλέπουμε ότι δεν ισχύει. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν οργανισμοί και φορείς οι οποίοι προσδίδουν μεγάλη σημασία στην ιατρική περίθαλψη των φτωχών ή των αστέγων. Αλλά από πλευράς ιατρικών υπηρεσιών και προγραμμάτων βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μία ολοκληρωμένη πολιτική. Γι' αυτό Πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να οριστεί εκ νέου, έτσι ώστε να υπάρχει ιατρική περίθαλψη, πλήρης ιατρική περίθαλψη και για τους άστεγους. Ευχαριστούμε τον κύριο Τανασέσκου. Επίτροπος έχει το λόγο για να κλείσει, να προσπαθήσει να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη δείχνει ένα έλλειμμα αλληλεγγύης και μέχρι ότου αυτή η κατάσταση αντιστραφεί όχι μόνο μπορεί να καταστρέψει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο αλλά και την Ευρωπαϊκή την Ένωση την ίδια. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Χωρίς πολύ ισχυρότερη αλληλεγγύη δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Και είναι αλήθεια ότι ενώσο γίνεται αυτή η μάλλον η κρίση, οι, τα κάτι μελη αλλά και οι περιφέρειές τους θα συνεχίσουν να οδηγούνται σε κοινωνική κρίση και κοινωνική καταστροφή ενδεχομένως και η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα στοιχεία αυτής της πολύ αρνητικής τάσης. Εγώ είμαι ευγνώμων στους βουλευτές γιατί αυτή η συζήτηση επιβεβαιώνει πως το σώμα είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει την έλλειψη στέγης και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η στρατηγική 2020 για την αντιμετώπιση της, της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού καταπολεμεί τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη και, και την παρουσία των αστέγων. Δεν οφείλεται αυτό στην έλλειψη στέγης, στην έλλειψη κατοικιών. Οφείλεται στην ε, παρακμή του πληθυσμού. Δεν πρόκειται για έλλειψη κατοικιών λοιπόν. Ε, και θα είναι λάθος να θεωρούμε τους στοχούς ε, και τους αστέγους ως ε, εγκληματίες. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών και οι τοπικές αρχές θα πρέπει να παρέμβουν για να διορθώσουν αυτήν την πολύ σημαντική αποτυχία. Οι άστεγη και η αντιμετώπιση της στόχιας είναι αρμοδιότητα του των κρατών μελών και ορισμένα κάτι μέλη ε, τη, ε, θεωρούν απόλυτα δική τους αρμοδιότητα. Ε, αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι περισσότερο συντονισμό των πολιτικών, όπως ε, τόνισε και η Λίζ Λίν, η ανταλλαγή των στατιστικών πληροφοριών και καλύτερη ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών. Ωστόσο, η Κομισιόν έχει ήδη ξεκινήσει δουλειά πάνω στις γραμμές που προτάθηκαν όπως για παράδειγμα έχει αρχίσει να βελτιώνει την γνώση, την καινοτομία και πιστεύω πως ε, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε πιο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και θα ήθελα να ανοίξω την πόρτα από τη νέα ομπρέλα της κοινωνικής καινοτομίας. Το πρόβλημα επίσης συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έλλειψη του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε από διάφορες πτυχές και από την νομοθετική. Γιατί αλήθεια είναι απαράδεκτο αν για παράδειγμα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ε, κόσμος που πήρε ένα δάνειο ε, υπόθηκο δάνειο χάνει το σπίτι του και το διαμέρισμά του και εξακολουθεί να χρωστά χρήματα στην τράπεζα. Ενώ έχει μείνει άστεγο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Επιπλέον η Κομισιόν είναι σε διάλογο με του ε, φορεί για να εξασφαλίσει ότι θα... το νομικό πλαίσιο θα είναι κατάλληλο. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε τη συνεργασία με τα κρατημέλη, ορισμένα από αυτά αντί να δουλέψουν για στρατηγική κοινωνική κατοικία, ανοίγουν το δρόμο για την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος. Στην Κρακοβία τον, τον, τον Οκτώβριο στην διάσκεψη για την ε, φτώχεια, για την πλατφόρμα για τη φτώχεια, να συνεχίσω το διάλογο, να παροτρύνω τα κατημέλη όπως ζήτησαν τα, τα, οι βουλευτές, αλλά και τους ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να συνεργαστούν σε αυτό το τομέα. Επίσης συνεχίζουμε τη δουλειά και τη συνεργασία με τις ΜΚΟ. Όλοι γνωρίζετε βέβαια πως δεν συμμερίζονται όλοι οι ΜΚΟ την προσέγγιση της διάσκεψης συνένεσης. Σε αυτό το συνεχιζόμενο διάλογο βασίζομαι λοιπόν στη στήριξη του σώματος αυτού για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αστέγων και να βελτιώσουμε τις συνθήκες στέγασης σε ολόκληρη την Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ε, έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και έχει κατατεθεί σχετικό ψήφισμα. Και περνάμε τώρα στην επόμενη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Καλώς ορίσατε κυρία Εντεγκάρντ.